Καλημέρα αγαπητοί συνάδελφοι. Επαναλαμβάνεται η συνεδρία στα πρακτικά της χθεσινής συνεδρίασης και τα κείμενα που έχουν εγκριθεί είναι στη διάθεσή σας. Υπάρχουν αντιρρήσεις. Όχι. Οπότε τα πρακτικά εγκρίνονται. Περνάμε στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης. Συζήτηση για ένα επίγον θέμα σύμφωνα με το άρθρο 162 του κανονισμού ανάμειξη άλλων χωρών στις δημοκρατίες μας και τις εκλογές μας. Θα ήθελα να σου πω ότι εδώ πέρα δεν θα επιτραπεί η διαδικασία του KHDI, ούτε θα γίνουν δεκτές μπλε κάρτες. Δίνω λοιπόν πρώτα τον λόγο στην ε, εισηγήτρια από την ομάδα Renew Europe για τέσσερα λεπτά. Αγαπητοί συνάδελφοι, τα τελευταία χρόνια έχουμε δει μια τεράστια αλλαγή στο πώς ε, διεξάγονται οι εκλογές. Έχουμε ακόμα φυλάδια, χτυπάμε τις πόρτες, ε, κάνουμε συζητήσεις στην τηλεόραση, αλλά οι ψηφοφόροι μας λαμβάνουν τις πληροφορίες τους από το διαδίκτυο, από τα κοινωνικά μέσα και τις στοχευμένες διαφημίσεις διαφημίσεις οι οποίες εκμεταλλεύονται όλο και πιο αποτελεσματικούς αλγόριθμους που στοχεύουν πλέον ατομικά. Οι πολίτες ε, σε ολόκληρη την Ευρώπη είναι στο έλεος του οποιοδήποτε έχει έναν υπολογιστή και ένα στόχο που θέλει να πετύχει. Έχουμε λοιπόν κοσμογονικές αλλαγές ε, που είναι σοβαρότερες ε, από την τυπογραφία, το ραδιόφωνο και την τηλεόραση. Το κενό όμω μεταξύ τη νομοθεσία αυτή αφενό και της ε, νομοθεσία και ρυθμίση ε, αφετέρου έχει γίνει πλέον πολύ μεγάλο και κυριολεκτικά και μεταφορικά οι παλιοί κανόνε δεν ισχύουν καθώ η νομοθεσία μα έχει μείνει πολύ πιο πίσω από την πραγματικότητα. Η άρνηση των εταιριών όπω το Facebook να αναλάβουν αποφασιστική δράση για να αστυνομεύσουν την ε, πλατφόρμα ανοίγει μια πόρτα στις εκλογές από την οποία μπορεί να περάσει οποιαδήποτε ξένη δύναμη. Η σωστή ρύθμιση πλατφορμών όπως το Facebook δεν παραβιάζει την ελευθερία του λόγου. Είναι το ηθικό μας καθήκον. Πρέπει να αναλάβουμε σοβαρότερη δράση κατά των ψεύτικων προφίλ και λογαριασμών. Να ενταθεί η προσπάθειά μας κατά της παραπληροφόρησης και η εκλογική νομοθεσία να έρθει στη σύγχρονη εποχή. Πρέπει να ερευνήσουμε τη χρηματοδότηση πολιτικών κομμάτων από το Κρεμλίνο. Παραδείγματο χάρη στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ξέρουμε ότι οι Ρώσοι ολιγάρχε έχουν δώσει πάρα πολλά λεφτά για να παίξουν τέννη με τον Μπόρι Τζόνσον. Εχθρικέ κυβερνήσει εκμεταλλεύονται τον ψηφιακό χώρο για να παρέμβουν στι εκλογέ μα. Με του δικού του στόχου. Έχουμε 50 εκλογικέ αναμετρήσει στην Ευρώπη μέχρι το 2020. Πρέπει λοιπόν να αρχίσουμε να το παίρνουμε στα σοβαρά. Αυτοί οι οποίοι μισούν την δημοκρατία και θεωρούν ότι οι εκλογές είναι απλά ένα πανηγύρι ε, μεταξύ των οποίων ε, και ο Βλαδίμιρος ε, Πούτιν ρίχνουν εκατομμύρια για να τις στρεβλώσουν. Τα έχουμε δει αυτά στην Ισπανία και στο Ηνωμένο Βασίλειο και στην Ιταλία. Αλλά δεν είναι μόνο ο Πούτιν. Γνωρίζουμε ότι ο Ντόμινικ Κάμιγκς, σύμβουλος του Πρωθυπουργού μας, είχε περάσει κάποιο καιρό στη Ρωσία. Αυτό πρέπει να ερευνηθεί. Και πολλοί εδώ πέρα βρίσκονται Εξαιτία του Steve Bannon. Και βεβαίω, ε, πολλοί δέχονται ευχαριστώ την βοήθεια των εξωτερικών δυνάμεων για να αναλάβουν την εξουσία. Θα κοίταγα προ τον κύριο Φάρατζ, αλλά δεν ήρθε αυτή την εβδομάδα. Επίση, απευθύνομαι προ τον Πρωθυπουργό του Ηνωμένου Βασιλείου που έχει αρνηθεί να δημοσιεύσει μια έκθεση του Κοινοβουλίου για τι παρεμβάσει τη Ρωσία στο δημοψήφισμα για τον Brexit του 2016. Εμεί όμω ξέρουμε τι γράφει αυτή η έκθεση, αλλά δεν την δημοσιεύει γιατί η αλήθεια μπαίνει εμπόδιο στις προσωπικές του φιλοδοξίες. Ο Μπόρις Τζόνσον πρέπει τώρα να δημοσιεύσει την έκθεση για τη Ρωσία. Τα πράγματα πλέον είναι τόσο άσχημα, ώστε η κυβέρνηση παριστάνει ότι έχει ένα site το οποίο ελέγχει ποιες ειδήσει είναι έγκυρες. Ο Βλαδίμηρος δεν χρειάζεται πια να κάνει τίποτα έχει εδρεωθεί πλέον η εκλογική παρέμβαση ξένων δυνάμεων και έχει γίνει ο κανόνα. Πρέπει να υπάρξει μια κοινοβουλευτική απάντηση σε αυτή την απαράδεκτη συμπεριφορά και αποφασιστική δράση στα κράτη-μέλη και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κι όμω οι πολιτικοί μέχρι στιγμή δεν κάνουν τίποτα. Το Facebook εξακολουθεί να λειτουργεί ω δούριο ύπο στη δημοκρατία μα. Έχει φτάσει η στιγμή το νέο αυτό κοινοβούλιο, η νέα αυτή κομισιόν να σοβαρευτούν. Αλλιώ θα είμαστε πάντα στο έλεος οποιοδήποτε αυταρχικού έχει ένα πληκτρολόγιο. Ελπίζω να συμμερίζετε κι εσείς αυτή την αίσθηση κινδύνου. Thank you very Ευχαριστώ. Να παρακαλέσω τους συναδέλφους, αν θέλουν να συζητήσουν, να μην γυρνάνε την πλάτη τους ε, στο Προεδρείο και ας καθίσουν... Ναι, σας παρακαλώ. Ου, Γεια σας. Ε, γιατί ακούγεστε. Δεν θα με ακούγατε δηλαδή χωρίς μικρόφωνο. Ευχαριστώ. Ε, καθίστε ο ένας δίπλα στον άλλον και μιλάτε χαμηλόφωνα. Θα δώσω τώρα τον λόγο στην Υπουργό την κυρία Τουπουράινεν. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αξιότιμη Ευρωβουλευτέ. Ο, ο Τζεφ Κέννιντ είπε κάποια στιγμή ότι μερικές φορές α, ε, ακόμη και οι ενωθεί μια ψήφου στην δημοκρατία ε, αποβαίνει βάρο του συνόλου τη κοινωνία. Οπότε η εξωτερική παρέμβαση σε εκλογικέ διαδικασίε έχει παρόμοιου κινδύνου στην κοινωνία. Κακόβουλε τέτοιε παρεμβάσει και χειραγώγηση διαδικτυακή ε, θέτει σε κίνδυνο τους δημοκρατικούς μας θεσμούς. Ε, αυτός ο κίνδυνος είναι πραγματικός και χρήζει άμεσης προσοχής. Χαίρομαι για την ευκαιρία που μας δίνετε να συζητήσουμε αυτό το τόσο σημαντικό ζήτημα σήμερα. Επαναλαμβάνω, η Φιλανδική Προεδρία έχει ως προτεραιότητα να συνεχίσει προσπάθειες και να ευαισθητοποιήσει την κοινωνία, να αυξήσει την ετοιμότητα και να ενισχύσει την αθεκτικότητα των δημοκρατιών μας απέναντι στην παραπληροφόρηση. Οι υβριδικές απειλές και η εξωτερική παρέμβαση στις δημοκρατίες μας εξακολουθεί να είναι ύψτη προτεραιότητα του πολιτικού μας προγράμματος. Η Προεδρία έχει λάβει ε, σειρά, έχει ε, αναλάβει σειρά προσπαθειών για παράδειγμα, έχουμε μια οριζόντια ομάδα εργασία του Συμβουλίου που δημιουργήθηκε κατά τον πρώτο μήνα ανάληψη Φιλανδική Προεδρία. Η ομάδα αυτή εργασία ε, εξετάζει την ενίσχυση τη ικανότητα Ευρωπαϊκή Ευρωπαϊκής ε, Ένωση να αντιταχθεί σε υβριδικέ απειλέ και να ενισχύσει την ανθεκτικότητα των κρατών μελών. Η εντολή τη ομάδα αυτή περιλαμβάνει και εξτρατή παραπληροφόρηση και παρέμβαση σε εκλογικέ διαδικασίε. Και μάλιστα προτείναμε ε, τις, τα συμπεράσματα του Συμβουλίου για το Δεκέμβριο για συμπληρωματικέ προσπάθειε να ενισχύσει αντιμετωπίσουμε την ανθεκτικότητα και να αντιμετωπίσουμε τέτοιε υβεριδικέ απειλέ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα συμπεράσματα αυτά στόχο έχουν και την καταπολέμηση τη παραπληροφόρηση για την εξασφάλιση ελεύθερων και δίκαιων εκλογών. Κυρία Πρόεδρε, αξιότιμοι Ευρωβουλευτέ, στη τελευταία συζήτηση που έγινε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, το Σεπτέμβριο ε, κατέληξε σε συνένεση ότι η παραπληροφόρηση και αυτές οι υβριδικές απειλές δημιουργούν κίνδυνο στη δημοκρατία και στις ευρωπαϊκές αξίες. Αναμφίβολα, τα κοινοτικά θεσμικά όργανα και τα κράτη-μέλη θα πρέπει να διαδραματίσουν πολύ σημαντικό ρόλο στα πλαίσια της εντολής και των αρμοδιοτήτων της προκειμένου να περιφρουρήσουν και να διαφυλάξουν τις δημοκρατίες τους. Η προστασία της ευρωπαϊκής